Με βάση την ε, ημέρησια διάταξη θα ακούσουμε τη δήλωση ε, Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους κανόνες για το ΦΠΑ και την ενιαία θηρίδα για το ΦΠΑ για τις ψυχιακές υπηρεσίες, ε, βιβλία και έγγραφα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος Άντσιπ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει τη δήλωση. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, θα ήθελα να σας δηλώσω ότι η Κομισιόν